Καλησπέρα σας. Τώρα είναι η ώρα των επεξηγήσεων ψήφου και πρώτη είναι η κυρία Μακοβέη. Ουσβεκιστάν, Εξήγηση Επεξήγηση ψήφου για την έκθεση τη σύσταση τη κυρία Μαρία Αρένα για την συμφωνία εταιρική σχέση με το Ουσμπεκιστάν.